Συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Έχει θέσει πίσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, λυπούμε για την καθυστέρηση με την οποία αρχίζουμε. γιατί η συνεδρίαση των συντονιστών κράτησε παραπάνω από ό,τι νομίζαμε. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να καθίσετε. Αρχίζει η συνεδρίαση. Παρακαλώ, συγχωρήστε μα για την καθυστέρηση με την οποία τελείωσε η συνάντηση των συντονιστών. Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να σα πω τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση των κανονισμών. Κύριο Σταρά ορίστηκε εισηγητή για την έκθεση πρωτοβουλία από κοινού με την υποεπιτροπή ΣΕΝΤ για την χρηματοδότηση της ε, πολιτικής ασφαλείας και για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και την σχετική έκθεση με τα δύο τμήματα Άνοιξη και Φθινόπορο η Γκούε θα μας προτείνει η συγητή. Για τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού 1150 του 2000 για τους ιδίους πόρους θα επανέλθουμε σε λίγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε μπει στη φάση μετά την συνδιαλλαγή χωρίς συμφωνία. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους <coughs> για, τον, για την αυστηρότητα με την οποία ακολουθήσαμε αυτά που είχαμε καθορίσει. Τη στρατηγική μας δηλαδή προσέγγιση με σαφές όραμα <clears throat> για τον προπολογισμό και τις γενικές του προτεραιότητες υπέρ της απασχόλησης, της καινοτομίας, της ανάπτυξης, αλλά επίσης και με την υποχρέωση να αντιμετωπίσει η Ένωση και τις υποχρεώσεις που έχει πληρωμών. Δυστυχώς υπάρχουν, έχουν έρθει στην Κομισιόν λογαριασμοί που πρέπει να τους πληρώσουμε και εδώ και πέντε χρόνια η χιονοστιβάδα αυτή συνεχώς αυξάνεται και πρέπει κάποτε να τελειώσουν όλα αυτά. Το 2014 ήδη φέτος δηλαδή από τον διορθωτικό προϋπολογισμό χρειάστηκαν ακριβώς έκτακτα μέτρα για να πληρωθούν τα πρόστιμα και ζήτησε η Κομισιόν να μεταφέρει στα κράτη-μέλη την ευθύνη αυτή. Εμείς δεν συμφωνούσαμε και χρειάστηκε να εξηγήσουμε στους εκλογείς μας τι κάνουμε δημοσιονομικά. Εδώ και τρεις εβδομάδες είχαμε προενώπιόν μας ένα συμβούλιο που περιοριζόταν να λέει ότι η συνδιαλλαγή έπαθε ημιπληγία γιατί λειτουργούσε λέει μόνο το ένα τμήμα του εγκεφάλου και το άλλο ήταν νεκρό. Και χρειάστηκε να φτάσει το μεσημέρι της 21ης μέρας για να καταλήξουμε ότι είναι απαράδεκτη η συνδιαλλαγή. Απαράδεκτη διότι το ύψος των πληρωμών δεν αρκούσε, δεν συμφωνούσε με τις προσδοκίες μας, 2 δισεκατομμύρια το 14 και 800 εκατομμύρια για το 15 Σύνολο σας υπενθυμίζω ότι για την περίοδο 14 <clears throat> με 15 <clears throat> χρειαζόμασταν 7 πρόσθετα δισεκατομμύρια για τις πληρωμές και το Συμβούλιο μας πρότεινε 3. 3.200. Και το απόγευμα ή προς το βραδάκι πρότεινε η Κομισιόν μία ενδιάμεση λύση τα 3,8 από τα 3,8 τα μισά, 1,9 δηλαδή, να διατεθούν και οι υφυπουργοί. Ο υφυπουργό Οικονομικών της Ιταλικής Κυβέρνησης που είχε την Προεδρία μαζί με ορισμένους άλλους πρεσβευτές και δημοσιονομικούς συμβούλους τα συζήτησαν όλα αυτά. Επί τρεις εβδομάδες δεν μπορούμε να πούμε ότι σεβάστηκαν τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου. Δεν ήρθαν υπουργοί πλήρης και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, σε λίγο θα μας στέλνουν μόνο βοηθούς στη συνδιαλλαγή. Πρέπει λοιπόν να γίνει σεβαστό το κοινοβούλιο και πρόκειται για την πρώτη συνδιαλλαγή μετά τις ευρωεκλογέ. Και δεν μας σεβάστηκαν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Το πρωί συνάντησα την κυρία Γεωργίεβα και συζητήσαμε τι χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να εγκριθεί ίσως το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015 και η διορθωτική προϋπολογισμή του 2014 κατά την Ολομέλεια στο Στρασβούργο την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Θα ήθελα λοιπόν να σας αναφέρω αυτό το πιθανό χρονοδιάγραμμα. Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι σε θέση να αποφασίσει την επόμενη Παρασκευή στις 28 Νοεμβρίου. Το σημαντικό όμως είναι ότι στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και πανενωσιακός, δηλαδή σε επίπεδο Προεδρίας της Κομισιόν, Προεδρίας του Κοινοβουλίου, Προεδρίας του Συμβουλίου, πρέπει να βρεθούν συμβιβασμοί και λύσεις σαφείς με όλα αυτά τα όργανα, όχι με απουσία του Κοινοβουλίου. Πρέπει το Συμβούλιο λοιπόν να μας πει καθαρά τι πρεσβεύει για τις πληρωμές. Επίσης τα ειδικά όργανα και εργαλεία πρέπει και μέσα πρέπει να βγουν από τα ανώτατα όρια να εξαιρεθούν. Για μας είναι κόκκινη γραμμή αυτό. Και η Επίτροπος θέλει να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να βγούμε από την ασάφεια. Να μην περιμένουμε την επόμενη ευκαιρία συνδιαλλαγής. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες για τις πληρωμές. Ως προς τις πληρωμές λοιπόν θα έπρεπε να πούμε ότι για να πληρωθούν οι πιο επίγουσες πιο επίγοντες λογαριασμοί που μας έχουν στείλει. Πρώτον, να δοθούν εξαιρετικώς ποσά για την πληρωμή των παλαιών λογαριασμών. Δύο, να ζητήσουμε για αυτό το θέμα των χρεών που έχουμε το Συμβούλιο να αναλάβει τη δέσμευση να πληρώσει τα χρέη αυτά. Δεν μπορούμε χρόνο με το χρόνο να συνεχίζουμε απλώς να παραπονούμαστε γιατί υπάρχουν απλήρωτοι λογαριασμοί. Τουλάχιστον η Κομισιόν είναι σαφής. Είναι πολύ δυσάρεστο να αρχίζει κανείς μια συζήτηση με την πρόταση της Κομισιόν για 7 δισεκατομμύρια και τελικά στη συνέχεια να μας λέει ε, μπορούμε και με λιγότερα. Εμείς ζητούμε από την Κομισιόν να προγραμματίσει τις πληρωμές που χρειαζόμαστε. Γιατί υποθέτουμε ότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας ορισμένων, μαξιλαράκια δηλαδή, και επομένως πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει με αυτές τις λεγόμενες outstanding payments, εκρεμείς λογαριασμούς και πρέπει ρητά να πούμε ότι τα ειδικά εργαλεία ευελιξίας θα εξαιρούνται, θα είναι έξω από τα ανώτατα όρια. Αν αυτά τα δεχτούν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο συμφωνίας όπως σας είπα μπορεί και να βρεθεί λύση. Την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ίσως γίνει μια πρώτη συνάντηση συντονιστών με την Επίτροπο για έναν απολογισμό που βρίσκονται οι συζητήσεις δηλαδή. Και η Επίτροπος μας είπε ότι μπορεί η Κομισιόν να δεχτεί στις 28 είπε Νοεμβρίου το σχέδιο προπολογισμού. Ότι αυτά συνθήκας λοιπόν πρώτος τριμερής διάλογος μπορεί να γίνει στις 2 Δεκεμβρίου. Ίσως προηγουμένως να γίνει και μια συνεδρίαση στην Επιτροπή μας αλλά δεν ξέρω αν θα χρειάζεται για να ούτως ή άλλως οι συντονιστές θα τα συζητήσουν και η Κομισιόν θα συνεδριάσει στις 3 4 Δεκεμβρίου και ίσως να γίνει τριμερής διάλογος να αρχίσει στις 8 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Προϋπολογισμών, η δική μας δηλαδή, στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει για να επικυρώσει το σχέδιο προϋπολογισμού. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες διότι φανταζόμαστε ότι η Κομισιόν στην προστασία του προϋπολογισμού θα τη συμπεριλάβει τις δικές μας τροπολογίες που εγκρίναμε στην προηγούμενη Ολομέλεια. Ε, λοιπόν, το Συμβούλιο ίσως να δεχτεί το σχέδιο προϋπολογισμού στις 15 Δεκεμβρίου και το ίδιο βράδυ θα συναντηθούμε εκτάκτος στο Στρασβούργο το βράδυ είπε για να εγκρίνουμε επίσημα το σχέδιο προϋπολογισμού και να επικυρώσουμε τη συμφωνία μας με τις τροπολογίες έτσι ώστε στην Ολομέλεια 17 Δεκεμβρίου με ψηφοφορία να μπορέσουμε να εκφράσουμε την έγκρισή μας του προϋπολογισμού 2015. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε, θελήσαμε να χειριστούμε τα πράγματα και τη συνένεση που σημειώθηκε και δεν μειώθηκε καθόλου καθόλου την διαπραγμάτευση, της συνδιαλλαγή. Θα έπρεπε λοιπόν να καταλήξουμε σε επιτυχία λόγω αυτής της τάσης, καταλήξαμε σε αποτυχία, τουλάχιστον δηλώσαμε ρητά τι θέλαμε και πρέπει αυτό να το ξέρουν και οι συμπολίτες μας. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν, μετά την αποτυχία αυτή της συνδιαλλαγής, πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο για να διατηρήσουμε αυτή την ομοφωνία ή συνένεση στο Κοινοβούλιο γιατί τότε είμαστε ισχυρότεροι. Κυρία Καζαμπάν. Ευχαριστώ πολύ. Συνοψίσατε τέλεια την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή και ποια είναι τα επόμενα βήματα τουλάχιστον ε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αξιολόγηση αυτή τη ε, διαδικασία συνδιαλλαγή, διότι πάντα λέμε ότι δεν λειτουργούν τόσο καλά οι διαδικασίε συνδιαλλαγέ. Πάντοτε λέμε ότι ακριβώς ε, λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένο το Συμβούλιο έχουν πολύ περισσότερο πρόβλημα από εμάς να καταλήξουν μεταξύ τους σε συμφωνία. Αλλά Πιστεύω ότι στις διαδικασίες κατάρτισης προπολογισμού είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή την τελευταία στιγμή στο παραπέντε που λύγει προθεσμία δεν υπάρχει καν ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο για να υπερασπιστεί μια πρόταση επί της οποίας θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Αυτό έγινε αυτή τη φορά. Και γι' αυτό αυτές τις 21 ημέρες δεν σημείωσαν καμία πρόοδο, δεν υπήρξε καμία προσέγγιση στις θέσεις Κοινοβουλίου Συμβουλίου την τελευταία φορά, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο που είχε αποτύχει η συνδιαλλαγή, είχαμε παρόλα αυτά σημειώσει πρόοδο κατά το 90% των συμφωνίων που είχαμε και έμενε ένα μικρό μέρος ε, για το οποίο δεν υπήρχε συμφωνία και θα ήταν εύκολο να συμφωνήσουμε. Και πράγματι το καταφέραμε και δεν χρειάστηκε να μπούμε στα 12 τιμόρια. Τώρα όμως είμαστε στην αρχή ακόμα. Ο καθένας περιχαρακωμένος στις γενικές του γραμμές. Εμείς στηρίζουμε τις πληρωμές, είναι προτεραιότητά μας, παρά τις προτάσεις όμως της Κομισιόν, που έχει κάνει δύο ήδη προτάσεις τις τελευταίες μέρες, δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες. Δεν καταφέραμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Υπήρχαν πολλά στοιχεία των προτάσεων της Κομισιόν που θα έπρεπε να τα αξιολογήσουμε ένα προς ένα. Αφού δεν συμφωνούσαμε όμως στα νούμερα τα γενικά, γιατί να μπούμε στις λεπτομέρειες. Χρόνο έχουμε. Μέχρι την Ολομέλη του Δεκεμβρίου έχουμε χρόνο για να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά θα εξαρτηθούν τα πάντα. Από το πρώτον, κατά πόσον το Συμβούλιο θα συνεχίσει και θα προοδεύσει στις εσωτερικές διαπραγματεύσει, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε κάπου στη μέση. Θέλω να πω κάτι και να το ξεκαθαρίσω. Το Κοινοβούλιο θέλει συμφωνία επί του προπολογισμού. Και νομίζω ότι αυτό το λέμε και το έχουμε γράψει αν θέλετε. Θέλουμε ένα προϋπολογισμό. Όχι όμως με κάθε τίμημα. Και γι' αυτό είμαστε και πάρα πολύ σταθεροί και εμένουμε στις θέσεις μας. Όχι βέβαια με άκαμπτο τρόπο. Έχουμε μετακινηθεί πάρα πολύ σε σχέση με την αρχική μας θέση μέχρι τις θέσεις της Κομισιόν. Εμείς όμως για να μπορέσουμε να προσυπογράψουμε μια συμφωνία πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάποια ελάχιστα επίπεδα που θέλουμε θα τα έχουμε για τις πληρωμές και τις προτεραιότητές μας, που δεν είναι και πολλές. Αλλά αφήσαμε κατά μέρος τους συμβιβασμούς, αφού δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Επρόκειτο για τους συμβιβασμούς που είχαν, κατά 99,9% που είχαν βάλει στο σχέδιο ε, κομισιόν δηλαδή. Βέβαια, δεν μας ικανοποιούσε απόλυτα ούτε πρόταση της Κομισιόν. Βρίσκαμε ανεπαρκή κάποια νούμερα, κάποια ποσά. Πώς βλέπω να βγαίνουμε από αυτό το αδιέξοδο, από αυτή την κατάσταση. Προφανώς οι επαφές μεταξύ Κοινοβουλίου και Προεδρίας του Συμβουλίου πρέπει να συνεχιστούν πιο έτσι, περιοδικά και να μην μένουμε μόνο σε τρεμερείς διαλόγους, δηλαδή να έχουμε πιο πολλές άτυπες ανεπίσημες συναντήσεις, κατηδίαν συναντήσεις, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε πιστεύω, να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια λύση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε. Ψάχνω τις λέξεις μου με προσοχή. Να είμαστε πιο χαλαροί με τα νούμερα λοιπόν. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά. Θέλουμε ένα σχέδιο πληρωμών, ένα πρόγραμμα πληρωμών. Αν είναι τόσο δύσκολη η θέση του Συμβουλίου και τόσο πολύ δυσκολεύονται να δώσουν κάποια στοιχεία αριθμητικά, κάποια ποσά κοντινά με αυτά τα οποία εμεί θεωρούμε απαραίτητα, η μόνη ε, περίπτωση να σώσουμε την κατάσταση είναι να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο Βέβαια έχοντας λάβει όλες τις πληροφορίες και έχοντας και τα, την τεχνική υποστήριξη της Κομισιόν πάνω σε ένα συγκεκριμένο πραγματικό πρόγραμμα πληρωμών, σχέδιο πληρωμών. Οι πληρωμές, οι λογαριασμοί είναι το θέμα. Πρέπει να πληρωθούν οι λογαριασμοί. Δεν μπορούμε να δεχθούμε όταν έχουμε απλήρωτους λογαριασμούς, ανεξόφλητους λογαριασμούς και ξέροντας ότι αυτό ζημιώνει πάρα πολύ κάποιες χώρες μέλη του Συμβουλίου. Δεν μπορεί να συσσωρεύονται λογαριασμοί απλήρωτοι. Αλλά στο Συμβούλιο τα έχουν βρει δύσκολα με τον προϋπολογισμό. Και εμείς τους θα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Και μιλώ και για τα κράτη-μέλη αυτά που έχουν λογαριασμού απλήρωτου και εμεί δεν του διευκολύνουμε για να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσει και η Κομισιόν να προγραμματίζει τις, ε, την πληρωμή των λογαριασμών. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο. Σα ευχαριστώ κυρία Γενική Συγγήτρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά του διορθωτικού προπολογισμού, η συγγητή μας είναι ο κύριο Ντεπρέ. Κύριε Ντεπρέ, έχετε εσεί το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ξέρω κι εγώ τώρα, χρειάζεται να πω κάτι. Είναι σαφή τα πράγματα πλέον. Το είπατε και επαναλάβετε επανειλημμένως. Αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε είναι το Συμβούλιο να συμφωνήσει με την πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 3, με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3 της Κομισιόν που ζητάμε επιπλέον κονδύλια της τάξης των 4,7 δις. 4,7 δις είναι ένα ποσό που μπορεί να αναπληρωθεί και με το παραπάνω από πρόστιμα, από καθυστερούμενους, από τόκους, από έσοδα δηλαδή ε, των κρατών. Δεν θα βγάλουν ε, από την τσέπη του. ούτε ένα ευρώ τα κράτη-μέλη για να πληρώσουν αυτά τα 4,2 δις. Απλά δεν θα βάλουν κι άλλα στην τσέπη του. Αυτό είναι το θέμα. Πού θα τα βάλουν, στα πορτοφόλια, στις τσάντες, στα όπου θέλετε, δηλαδή, στα, ε, τα παραπάνω αυτά έσοδα. Και δεν σέβονται τους κανόνες της αστερικής αγοράς, ε, δεσπόζουσα θέση και τα λοιπά, αυτοί οι όμιλοι που δεν τα σέβονται όλα αυτά πληρώνουν πρόστιμα και αυτά θα τα βάλουν στην τσέπη τους τα κράτη-μέλη. Εμείς θέλαμε αυτά τα λεφτά να καλύψουν τα κενά. Το Συμβούλιο θέλουμε να συμφωνήσει επί των ποσών που εμείς θεωρούμε απαραίτητα. Γιατί όπως πάντα είπαμε και έχουμε επενθυμίσει επανειλημμένο στην Επιτροπή αυτή Προπολογισμών, εάν εμείς αποδίδουμε τόσο μεγάλη σημασία. Σε αυτά τα επιπλέον κονδύλια για το 2014, σε αυτούς τους διορθωτικούς προπολογισμού. Γιατί το κάνουμε, ακριβώς γιατί είναι απαραίτητα τα κονδύλια αυτά, ώστε ο προπολογισμό του 2015 να μπορέσει να λειτουργεί σωστά, να έχει ένα νόημα αυτός ο προϋπολογισμός. Αλλιώς ξεκινάμε το 2015 με επιπλέον 5 δις χρωστούμενα. Άρα για μια ακόμη φορά δεν θα φτάσουν τα κονδύλια για το οικονομικό έτος 2015 και θα έχουμε νέα υποβάθμιση και θα έχουμε μεγαλύτερους ε, απλήρωτους λογαριασμούς. 23 δις είναι τώρα, θα γίνουν 28, ε, ίσως και 30 τα δις των ε, ανεξόφλητων λογαριασμών. Άρα αυτό θα μας οδηγήσει κάποια χρονική στιγμή σε μείζωνα αδυναμία πληρωμών, σε πλήρες αντιέξοδο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εμείς είπαμε ότι πρώτα-πρώτα θέλουμε συμφωνία για τους διαθετικούς υπερβολισμούς του 2014 και εσείς και εμείς τα κράτη-μέλη κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους πείσουμε να κάνουν αυτή τη χειρονομία, γιατί είναι προς όφελος όλων. Αφού δεν χρειάζεται να βγάλετε λεφτά από την τσέπη σας, τους λέμε. Θα το δούμε και στο επόμενο σημείο της Μεσιαδιάταξης. Το Συμβούλιο πάντως προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα του Κάμερον και έχει δαπανίσει πολύ πιο πολύ χρόνο για αυτό το θέμα παρά για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Παρότι είναι τόσο μεγάλες οι προκλήσεις και δικηβεύονται τόσο πολλά ε, με αυτό το θέμα και όχι με τον ε, καθόλου αξιοσέβαστο κατά τα λοιπά κύριο Κάμερον, που είναι και πολύ μικρά τα ποσά που του ζητάμε. Ευχαριστώ. Κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι κατανοούμε, όλοι προερχόμαστε από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανοούμε ότι είναι δύσκολο για το Συμβούλιο να καταλήξει σε μία θέση. Βλέπω και στις γερμανικές εφημερίδες τι διαστάσεις δίνει ο αρμόδιος υφυπουργός και μπορώ να κατανοήσω σε ποια κατάσταση βρίσκονται και οι χώρες μέλη. Αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να λύσουμε τα προβλήματα του Συμβουλίου Υπουργών και των χώρων μελών. Υπάρχουν βεβαίω περιορισμοί, υπάρχουν δυσκολίε με του εθνικού προπολογισμού. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμω παρόμοιοι περιορισμοί, δυσκολίε και στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Που ωστόσο το περιεχόμενό του καθορίζεται από τι εντολέ που δίνουν οι χώρε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα πράξει και τι θα παραλείψει. Επομένω, δεν μπορούμε να του απαλλάξουμε από τι υποχρεώσει του. Κατανοώ, όπω είπα, πάλι την κατάσταση των εθνικών δημοσίων οικονομικών, αλλά πώς θα είναι βιώσιμος στο μέλλον ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό Και δεν βλέπω την παραμικρή διάθεση από πλευρά χωρών μελών να λάβουν τι ευθύνε του. Ακούω όλο αυτό το μπλα μπλα για εξοικονομήσει και από την άλλη μεριά, αγαπητέ συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω όπου υπάρχουν συμφέροντα του Συμβουλίου να μην υφίσταται πλέον το δόγμα αυτό των εξοικονομήσεων, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου ο καθένας αναγνωρίζει ότι ο αριθμός των δικαστών είναι πλέον πολύ μικρός, είναι ανεπαρκής, δεν μπορεί το δικαστήριο να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του με τους υφιστάμενους 28 δικαστές. Και η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρόσφυγες για αποζημιώσεις για αποζημιώσεις επειδή ακριβώς καθυστερούν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και λέμε τώρα να αυξηθούν οι δικαστέ από 28 σε 40. Τι κάνει το Συμβούλιο, δεν μπορεί καν να συμφωνήσει από πού θα πάρει, από ποιε χώρε θα πάρει του 12 παραπάνω δικαστέ. Και η λύση, α, όχι 40, θα βάλουμε 56, ώστε η κάθε χώρα να έχει δύο δικαστέ. Κανένα πρόβλημα εκεί. Το πώ θα χρηματοδοτηθούν αυτοί, δεν είπε κανένα καμιά απάντηση. Επειδή πρόκειται για συμφέρον των χωρών μελών, ξαφνικά δεν του ενδιαφέρει η εξοικονόμηση. Ας προσλάβουμε άλλους 16 δικαστές. Με πικραίνει αυτή η κατάσταση, το λέω καθαρά, διότι ακούμε ξανά και ξανά από τις διάφορες χώρες μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περικόψει τις δαπάνες της. Πρώτο λοιπόν αυτό. Όπου σιγά σιγά πέρα από πίκρα αισθάνομαι και οργή για τις θέσεις του Συμβουλίου Υπουργών. Και όπως είπα, βλέπω καλά ποια είναι η θέση των ε, χωρών μελών που στην ουσία οδηγεί σε μια οργανωμένη από μέρους τους αδιαφορία. Τώρα έχω μια πρόταση για την παραπέρα πορεία των ε, διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρός μας τόνισε προλίγου ότι στο μέλλον θα στέλνουμε και εμείς τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς μας. Εγώ να κάνω μια λίγο διαφορετική πρόταση. Αν τα πράγματα είναι όπως έγιναν την προηγούμενη Δευτέρα, ότι απέναντί μας στο Συμβούλιο δεν κάθεται ούτε ένας που να έχει πραγματική εξουσιοδότηση να μπορεί να αντιδράσει στις προτάσεις της Κομισιόν, ε, τότε δεν χρειάζεται και εμείς να ασχολούμεθα. Αγαπώ την ε, εργασία μου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι μπορώ να κάθομαι κάπου εδώ και πολύ πιο βολικά στις Βρυξέλλες 9 η ώρα το βράδυ από ότι να είμαι εδώ στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω τους πρέσβεις να τηλεφωνούν στους αρμόδιους υφυπουργούς ή υπουργού του. και να υπάρχει θετική απάντηση από τον Υπουργό. Δεν έχω δει τέτοια πράγματα. Μόνο για να τους ενημερώνουν. Ε τότε ας κάνουμε το εξή. Ακούμε την άποψη του Συμβουλίου σκεφτόμαστε για λίγο αν μπορούμε να συμφωνήσουμε ή όχι, λέμε τη δική μας άποψη και σηκωνόμαστε και φεύγουμε, πάμε σπίτια μας. Και γλιτώνουμε και τα έξοδα, γλιτώνουμε και τους διερμηνείς και το χρόνο και την εργασία και τον κόπο και όλα αυτά. Μπορώ να τονίσω δηλαδή το εξή. Οι πληρωμές πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Οι εξοφλήσεις των απλήρωτων λογαριασμών. Μέχρι τώρα από το Συμβούλιο δεν βλέπω καμία πρόταση, ούτε καμία σταθεροποίηση της κατάστασης. Πολύ λιγότερο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ολόκληρο παλιροϊκό κύμα που έχουμε ανεξόφλητων λογαριασμών. Για να αρχίσουμε καν να λύνουμε το πρόβλημα. Δεν μας κάνουν καν προτάσεις για μια σταθεροποίηση. Και πώς θα λειτουργήσει χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τα ειδικά τα έκτακτα εργαλεία τα οποία είναι πάνω από τις όροφες. Δεν βλέπω τη λογική. Εάν δε το Συμβούλιο επεδείκνυε την ίδια προσοχή για το θέμα αυτό, όπως για, τις, για την υπόθεση που δίνει, την προσοχή μάλλον που δίνει στην υπόθεση των κάτω χωρών της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, που βέβαια έχουν και αυτές τις δυσκολίες τους, τότε θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ευχαριστώ. ο κύριο Φερνάντες. Έχω κύριε Πρόεδρε ορισμένε διαπιστώσεις και πρώτα το Κοινοβούλιο ήδη από την αρχή ήταν ενωμένο στο θέμα των ανεξόφλητων λογαριασμών. Δεύτερο, το Συμβούλιο αποδείχτηκε ότι δεν είναι ενωμένο στο ζήτημα του προϋπολογισμού συνολικά αλλά και βεβαίως για το σημαντικό πρόβλημα της πληρωμής των ανεξόφλητων λογαριασμών. Η ίδια πλειοψηφία στο Συμβούλιο που εγκρίνει προγράμματα, σχέδια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για νέους, για την έρευνα. Όταν έρθει η ώρα να πληρώσει, δεν εγκρίνει τις πληρωμές. Για τα έργα, για τα project εκείνα τα οποία ήδη είχε εγκρίνει να γίνουν. Διόλου δεν είναι το κοινοβούλιο που ζητάει δήθεν περισσότερα. Το κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί για να επιλύσει το πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών. Το μόνο που θέλουμε είναι να μην καταρρεύσει ο προπολογισμό. Το μόνο που θέλουμε είναι να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των θεσμών. Είναι σημαντικό να το κατανοήσουν αυτό όλοι και να συμβάλλουν όλοι. Όλα τα θεσμικά όργανα δηλαδή. Όχι μόνο το κοινοβούλιο. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να καταλήξουμε να λήξει το 2014 με 26 δισεκατομμύρια ανεξόφλητους λογαριασμούς. Υπάρχουν όμως χρήματα που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εν μέρη. Έχουμε 4,9 δισεκατομμύρια. Θα μας λείπουν λοιπόν 23. Το, κοινοβούλιο, το, Συμβούλιο εισπράττει χρήματα από, από πρόστιμα, από τόπους υπερημερίας, από το ένα από το άλλο. Να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά. Όχι. Θέλει αυτά να επιστρέψουν στα χρηματοκιβώτια των χωρών μελών. Κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι οι χώρες μέλη θα διαθέσουν 4,9 δισεκατομμύρια. Όχι, δεν είναι έτσι. Μιλούμε για όλα αυτά ότι το συνολικό και μόνο ποσό που θα πρέπει να καλύψει το ε, Συμβούλιο θα είναι 140 εκατομμύρια. Τίποτα δηλαδή άμα το διαιρέσεις δια 28. Ένα άλλο, σοβαρό πράγμα. Εμείς θέλουμε να δούμε να δημιουργείται ανάπτυξη, θέλουμε να δημιουργηθούν δουλειές. Έχουμε και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά τα πράγματα έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 14 έως 20, 2014 έως 20, δεν εφαρμόζεται καν. το 2014 είναι επιβαρημένο ακόμα από ανεξόφλητους λογαριασμούς προγραμμάτων του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε αναλάβει υποχρώσεις απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης όμως. Είπαμε θα φτιάξουμε, θα επενδύσουμε, θα επενδύσουμε στον αγώνα κατά της φτώχειας, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Πού είναι τα προγράμματα αυτά τα οποία υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί βέβαια η Επιτροπή να μην ζητήσει να γίνουν παραπάνω σχέδια. Αλλά είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή να προχωρήσει τι δραστηριότητε των προγραμμάτων που έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Κοινοβούλιο εν τέλει δεν ζητεί περισσότερα χρήματα από το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητούμε μοναχά οι υποσχέσει που έχουν δοθεί να τηρηθούν. Ο κύριος κύριε Πρόεδρε. θλιβερό το θεατρικό έργο που μας παίζουν. Αν ήταν τουλάχιστον καμιά κομμωδία θα γελούσαμε, αλλά είναι μάλλον δράμα. Σήμερα αναρωτιούνται οι πολίτες για την Ευρώπη και το μέλλον της. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Δεν έχουμε το δικαίωμα σήμερα να υποχωρήσουμε, να υπαναχωρήσουμε μπροστά στο Συμβούλιο. Γιατί αν το πράξουμε τότε θα ανοίξουμε την πόρτα σε όλους τους, θα στρώσουμε το δρόμο σε όλους τους ευρωσκεπτικιστές. Για τις πληρωμές πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέρμα, αλλιώς δεν θα επιδείξουμε πνεύμα υπευθυνότητας και ακόμα παραπάνω. Δεν πρέπει να παρατήσουμε καθόλου το θέμα και των δεσμεύσεων και των προβλέψεων που είναι ουσιώδεις και αυτές για το μέλλον. Αν δεν κάνουμε αυτή την προσπάθεια και για τις προβλέψεις, τότε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Και η Ευρώπη στο τέλος δεν θα έχει πια τα μέσα να ανταποκριθεί σε αυτά που δηλώνει για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τις υποδομές, για την ε, σύνδεση υψηλής ταχύτητας για τους νεολαία Πράγματα που τα λένε σε όλες τις χώρες, αλλά ακριβώς οι χώρες αυτές που λένε αυτά τα πράγματα αρνούνται να δώσουν τα μέσα, να μας δώσουν τα μέσα να εφαρμόσουμε τις δηλώσεις αυτές. Είναι σημαντικό να το θυμίζουμε αυτό και να προσέξουμε το θέμα και των δημοσιονομικών προβλέψεων όπως και των πληρωμών. Τώρα, καταλαβαίνει κανείς γιατί τα κράτη-μέλη που λέγονται καθαροί εισφορείς αντιδρούν. Όσο δεν βρίσκονται ευρωπαϊκοί πόροι και όχι εθνικοί, δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ας είμαστε λοιπόν πολύ στεναροί για τις πληρωμές, αλλά να μην ξεχνάμε και τις προβλέψεις για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτά που δηλώνουν η κυρία Ταπαρτέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν συμφωνώ με τους υπόλοιπους, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να καθοριστεί ρητά ότι η στάση του Συμβουλίου είναι πλήγμα στα θεμέλια της Ευρώπης. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη, πιστεύαμε ότι θα λυνόταν το πρόβλημα των πληρωμών αλλά βλέπουμε τώρα υπαλλήλους που δεν έχουν καν εντολή πολιτική να μη μας σέβονται. Πρέπει αυτό να σταματήσει. Έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες, το ίδιο επίπεδο ευθυνών, σε ισοτιμία με το Συμβούλιο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για τον προϋπολογισμό της Ένωσης ολόκληρης, όχι ειδικά του Κοινοβουλίου, τον οποίο πρέπει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο. Είμαστε λοιπόν σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν υπάρχουν πληρωμές προς τα κράτη-μέλη, δεν μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως όλα τα σχέδια και προγράμματα που έχουν αναλυφθεί και επομένως θα πληγεί έτσι και η οικονομία των εθνικών των χωρών μελών. Αυτό είναι ο φαύλος κύκλος, πρέπει να το πούμε αυτό και να προειδοποιήσουμε δηλώνοντας το ρητά στα κράτη-μέλη. Ίσως πρέπει να διατυπώσουμε μια επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί το πρόβλημα αυτό των καθυστερουμένων πληρωμών χρονίζει. Κάθε χρόνο το συζητάμε και δεν βρίσκουμε λύση. Ο προϋπολογισμός της Ένωσης στο κάτω-κάτω είναι ένα από τα θεμέλια της λειτουργίας της. Το πρόβλημα είναι λοιπόν σοβαρό. Ευχαριστώ κύριος Βιώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φυσικά συμφωνώ με αυτά που είπε πάτε και εσείς και ο συγχτής. Υπάρχει μεγάλη δυσφορία και μετά την αποτυχία της συνδιαλλαγής. Νομίζω τα είπαμε όλα, όλοι. Πριν λοιπόν προσπαθήσω να διατυπώσω μερικές συστάσεις, θα ήθελα να τονίσω τον κίνδυνο που υπάρχει και που τον ανέφεραν και άλλοι. Μπορεί, είναι πιθανό, να αυξηθούν τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα ορισμένων πολιτών Εκτός από το ότι δεν πληρώνουμε ορισμένους λογαριασμούς που χρωστάμε, υπάρχει και μεγάλη δυσαρέσκεια των πολιτών και δεν καταφέρνουμε να πείσουμε την κοινή γνώμη, να εξηγήσουμε τι είναι η δουλειά που κάνουμε όπως γίνεται κυρίως στην Ιταλία, ίσως στις άλλες χώρες ο τύπος να σέβεται λίγο περισσότερο τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά στην Ιταλία μερικές εφημερίδες λένε ότι οι ευρωβουλευτές περνάνε καλά και δεν κάνουν τίποτα και ζητούν από τα κράτη-μέλη 140 δισεκατομμύρια για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι λένε. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και να κάνουμε κάτι να εξηγήσουμε και στον τύπο περί τίνος πρόκειται. Το θέμα δεν είναι να πληρωθούν λογαριασμοί για τους καφέδες μας και τα ποτά μας, αλλά να πληρωθούν λογαριασμοί πολύ μηνύ. Δεύτερον. Ε, noi ora dobbiamo rimanere sicuramente uniti. Φυσικά πρέπει να συνεννοηθούμε με την Κομισιόν. Είναι φυσικό, ε, σίγουρο ότι πρέπει η συζήτηση να γίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και οι παρεμβάσεις μας να στοχεύουν σαφώς το προσδοκόμενο αποτέλεσμα και πέρα από αυτά πρέπει να ζητήσουμε η Ιταλική Προεδρία να παρέμβει και να μιλήσει με τρόπο σαφέστερο από ό,τι μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν εκτός από την μεγαλύτερη σαφήνεια να γίνουν όλα και πιο επίσημα και να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας επιτέλους. Δεν έχουμε πια το χρόνο για να καταστρώσουμε σχέδια στρατηγικής και τακτικής. Πρέπει όλοι μας <clears throat> που εκπροσωπούμε τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο δηλαδή, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει το Συμβούλιο να συζητήσει σοβαρά μαζί μας και με την Κομισιόν, σοβαρότερα. Να μην νομίζουμε ότι έχουμε όσο χρόνο θέλουμε. Και αυτή τη δουλειά να την κάνουμε την επεξηγηματική και στα κράτη-μέλη να το εξηγήσουμε και στους συναδέλφους μας, τους εθνικούς βουλευτές, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ότι πρέπει επιτέλους να ληφθεί μια απόφαση υπέρ του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Μόνκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, αλλά και τους εισηγητές και όλους τους συναδέλφους Πιστεύω ότι στις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετείχαμε δείξαμε ενότητα και η ενότητα είναι και η δύναμή μας. Δεν ισχύει το ίδιο το Συμβούλιο, ενώ έπρεπε να φαίνονται ή τα μπορεί να φαίνονταν εξωτερικά, δεν είναι ενωμένοι. Πιστεύω λοιπόν ότι αν επιμείνουμε θα πετύχουμε. Το Συμβούλιο δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του και αυτό δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε κάποια κράτη που είναι οι καθαροί εισφορείς. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον. Και σίγουρα αυτό δίνει όπλα στη φαρέτρα των ευρωσκεπτικιστών. Το θέμα είναι από πού θέλει να βρει τα χρήματα το Συμβούλιο. Μια πολύ επικίνδυνη εναλλακτική είναι κάποιοι από το Συμβούλιο να θελήσουν να αναβάλουν την ανανέωση κάποιων δεσμεύσεων, υποχρεώσεων, ανάληψεων υποχρεώσεων. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες εναλλακτικέ. Επαναλαμβάνω όμως ότι το Συμβούλιο δεν είναι ενωμένο, δεν έχει κοινή θέση. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε από κοινού με την Κομισιόν να πιέσουμε το Συμβούλιο και να το αναγκάσουμε να συμφωνήσει για μια διαφορετική μέθοδο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Άρα να μην εξαρτώμεθα από το κατά πόσο θα τηρεί τις δεσμεύσεις του ή το Συμβούλιο. Άρα θα πρέπει να βασιζόμαστε στους ίδιους πόρους. Να έχουμε ένα καλό σύστημα ιδιών Εκεί θα εστιάσουμε τη δουλειά μας στο μέλλον για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. και ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ας μην γίνεται σε εθνικό. Γιατί έτσι θα έχουμε και τη χρηματοδότηση που θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Merci, Madame. Ευχαριστώ η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να παραπέμψουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τρεις φορές τον προηγούμενο χρόνο αντιμετωπίσαμε παρόμοια κατάσταση. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν προσεκτικά πώς καταλήγουμε στην κατάσταση αυτή και πώς καταλήγουμε στην κατάσταση αυτή και είναι αντίθετη και με τη συνθήκη. Predsedujoči, hvala eh, eh, Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου ήθελα και εγώ να λάβω το λόγο στην συζήτηση που τη θεωρώ σημαντική. Εσείς προτείνατε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι πρόκειται να ξανασυναντηθούμε με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφενός αυτό το βρίσκω σωστό και εκεί πρέπει να βασιστούμε στα όσα ήδη έχουμε επιτύχει. Από την άλλη μεριά βρίσκω ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δυσχέρανση των ε, διαπραγματεύσεων. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε πλέον στην εφαρμογή των 12 τιμωρίων για το 2015. Μα τι μήνυμα είναι αυτό που θα δώσουμε τότε στους πολίτες μας που μας εξέλεξαν στο κάτω της γραφής για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αυτοί οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί οδηγούν σε μια, δίνουν μάλλον μια πολύ άσχημη εικόνα στον ενωσιακό προϋπολογισμό βρίσκω ότι λείπει η πειθαρχία. Πειθαρχία δηλαδή στην εξόφληση των λογαριασμών. Αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό και ιδίω αποθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αν έχω καταλάβει καλά, ανεξόφλητοι λογαριασμοί υπάρχουν ήδη από το 2010 και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Φοβούμαι ότι θα συνεχιστεί μάλιστα και του χρόνου. Και πέραν αυτό. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε, πώς θα καταφέρουμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο. Το Συμβούλιο Υπουργών οφείλει να μας δώσει επαρκείς πόρους ώστε να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τους λογαριασμούς. Αν δεν εγκριθεί έγκαιρα ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2014, σημαίνει αυτό ότι όλοι οι πόροι που πρόκειται για παράδειγμα από το Ταμείο Αλληλεγγύης και από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, όλα αυτά θα υποστούν μεγάλες περικοπές. Για τις 25 Νοεμβρίου βλέπω έχουν εγγραφεί όλες αυτές οι εκθέσεις. πρόκειται να εγκριθούν στην ημερήσια διάταξη. Αλλά αν κατάλαβα καλά, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν τότε να εξηγήσουμε στους ψυχοφόρους ότι δεν έχουμε χρήματα. Εδώ σημειώθηκαν στη Σλοβενία, τη χώρα μου, αλλά και στην Κροατία, πλημμύρες με τρομερές καταστροφές. Στην Ελλάδα σεισμοί. Πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό ότι δεν υπάρχουν πόροι για την αποζημίωση των ανθρώπων ή πάντως δεν θα αποζημιωθούν έγκαιρα. Έχουμε ξαναπεί ήδη εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι οι διαδικασίες για να απελευθερωθούν τα χρήματα αυτά, για παράδειγμα από το Ταμείο Προσαρμογής και Κοσμιοποίηση, είναι πολύ χρονοβόρες. Τώρα όμως, εμείς καθυστερούμε την αποπληρωμή, βεβαίως μαζί με το Συμβούλιο. Στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που προτείνατε για τις διαπραγματεύσεις, ελπίζω να μπορέσει να εξευρεθεί συνένεση, ώστε να εξοφληθούν και ανεξόφλητοι λογαριασμοί, αλλά και να μπορέσουν επίσης να καταβληθούν τα χρήματα των αποζημιώσεων στους πολίτες. Ωραία. Τελειώνει εδώ αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Το παράδοξο είναι ότι σε μερικές μέρες ο κύριος Γιούνκερ θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου του για τις επενδύσεις 300 δισεκατομμύριων και διάβαζα στον τύπο, στον Βρετανικό τύπο, τις δηλώσεις ενός Γάλλου Υπουργού που έλεγε ότι χρειάζεται φρέσκο χρήμα για αυτές τις επενδύσεις. Ενώ περί τίνος πρόκειται Έχουμε 30 δισεκατομμύρια απλήρωτους λογαριασμούς που δυσκολεύουν και τις επιχειρήσεις και άρα χειροτερεύουν και την κατάσταση της ανάπτυξης και της ε, καταπολέμησης της ανεργίας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε τις κυβερνήσεις ενώπιον των ευθυνών τους και ιδιαίτερα να μην αφήνουμε να λέγεται στις χώρες μέλη ότι είμαστε κοινοβούλιο που δαπανάει πολλά. Γιατί αφού έχουν αναλυφθεί οι δεσμεύσεις, όταν έρθει ο καιρός της πληρωμής πρέπει να γίνονται οι πληρωμές. Αυτό είναι το θέμα. Θα δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Γιούνκερ να μας πει τι έχει να πει για τον προϋπολογισμό και όχι απλώς να εκτελέσει τον προϋπολογισμό του κυρίου Μπαρόσο. Αλλά αναρωτιέμαι μήπως δεν θα έπρεπε να συνδέσουμε να βρούμε κάποια συνέργεια μεταξύ του προϋπολογισμού 15 και του σχεδίου επενδύσεων των 300 δισεκατομμύριων, γιατί αυτά τα 300 δισεκατομμύρια από πού θα προέλθουν. Από τη συλλογή της ιδιωτικής αποταμίευσης. Αλλά πώς θα φτάσουμε ως εκεί πρέπει να υπάρχει κάποια ελκυστικότητα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλει να κρατήσει το τριπλό αλφα της και όταν δημοσιεύει ομόλογα έργο τα κρίνει και η αγορά. Αλλά αυτό είναι μια μικροαπάτη γιατί η αγορά ξέρει ούτως ή άλλως αν θέλουμε να κάνουμε κάτι που δεν μπορεί να το πράξει η αγορά, χρειάζονται και εγγύησεις. Και τις εγγύησεις ποιος θα τις δώσει, τα κράτη-μέλη ή η ίδια η Ένωση. Ίσως πρέπει να κινητοποιηθούν και μερικοί πόροι που έχουν συσσωρευτεί στο Ταμείο Εγγυήσεων, Δημοσιονομικών Εγγυήσεων που δημιουργήθηκε ο, την εποχή της κρίσης των κρατικών χρεών στην Ελλάδα και αλλού ή να κινητοποιηθεί και ο μηχανισμός δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Θα δούμε. Πάντως πρέπει να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος που προ στιγμή δεν προβλέπεται. Δεν θα τα συζητήσουμε ξανά σήμερα για το πρόγραμμα των 300 δισεκατομμυρίων. Όλοι μας ελπίζουμε ότι δεν θα είναι απλώς μια απάτη αλλά και κάποια πραγματικότητα σας είπα ότι πρέπει το βασικό θέμα των πληρωμών των ειδικών εργαλείων να είναι εκτός των ανωτάτων ορίων και αυτό να συζητηθεί στο ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο. Να μην γίνεται κάθε χρόνο αυτή η διελκυστίνδα Συμβουλίου Κοινοβουλίου που μειώνει και την αξιοπιστία μας στα μάτια της κοινή γνώμης. Ζητούμε λοιπόν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να επιδείξουν συνέπεια και να πάψουν να στηρίζονται σε σημειώματα δημοσίων υπαλλήλων στα Υπουργεία που είναι βραχυπρόθεσμο οράματος και δεν λύνουν το πρόβλημα. Η Κομισιόν λοιπόν πράγματι μπορεί κάτι να κάνει, έχει περιθώρια. Αλλά στις επόμενες μέρες όταν θα επιστρέψετε στις χώρες σας και στις εκλογικές σας περιφέρειες. Σας ζητώ να πληροφορήσετε τις κυβερνήσεις σας, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι υπουργοί δεν τα ξέρουν όλα, και να κοινοποιήσετε, να... Ούτως ή άλλως εκείνη η γνώμη βέβαια δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα αυτά, αλλά να εξηγήσετε ότι υπάρχουν χρέη που συνεχώς αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, 5 δισεκατομμύρια το 10 και 30 σχεδόν σήμερα. Και ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Όταν υπάρχουν λοιπόν απρόβλεπτοι πόροι, γιατί πληρώνονται και πρόστιμα, πόσος χρόνος χρειάζεται για να δικάσει, εκδικάσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μία υπόθεση ανταγωνισμού. Τέσσερα χρόνια. Το 11 ζήτησαν οι δικαστέ τη δημιουργία 12 πρόσθετων θέσεων και μέσα σε τρία χρόνια δεν συμφώνησαν επ' αυτού τα κράτη-μέλη. Και το δικαστήριο είπε εμείς θα δημιουργήσουμε 28 θέσεις αφού είναι 28 οι χώρες μέλη και μετά μας λένε να μειώσουμε τις δαπάνες. Πώς. Απλό το μήνυμα λοιπόν. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τα χρέη της και όταν υπάρχουν απρόβλεπτοι πόροι πρέπει τα κράτη να αρνούνται να, τα βάλουν στην τσέπη, να τους βάλουν στην τσέπη τους για να καλοποιήσουν δήθεν τον προϋπολογισμό τους. Αυτά τα 30 δισεκατομμύρια χρεών πρέπει να προσθεθούν και στο έλλειμμα των κρατών μελών, που δεν είναι 30 δισεκατομμύρια, αλλά αν κάποια χώρα έχει κατά 15% συμβολή, στο χρέος αυτό προστίθεται και στο δικό της χρέος. Λοιπόν, μην αμφιβάλλετε για το αποτέλεσμα. Η θέλησή μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αλλά όχι όποια συμφωνία και να είναι. Αρχίζει η καινούργια θητεία και πρέπει να σεβαστούμε ορισμένες βασικές αρχές. Καταρχήν να γίνεται σεβαστό το κοινοβούλιο και έπειτα να γίνονται σεβαστές οι δεσμεύσεις μας. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να διατηρήσουμε την ενότητά μας μέχρι το τέλος γιατί το κοινοβούλιο μόνο ενωμένο είναι ισχυρό. Τώρα θα μιλήσουμε για την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού. Ξέρετε ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός 6 προβλέπει την πληρωμή 9 εκατομμυρίων από εισφορές των κρατών μελών με βάση ένα νέο ορισμό της προστιθέμενης αξίας και η Κομισιόν προτείνει 10 εκατομμύρια να κατανεμηθούν μεταξύ των χωρών μελών λιγότερα σε αυτούς που συνεισφέρουν λιγότερο στον προϋπολογισμό και περισσότερα οι άλλοι. Πάντως πρόκειται για επιστροφή σε εθνικό προϋπολογισμό. Η διαφορά μεταξύ 9,5 εκατομμυρίων και 10 είναι 500 πρόσθετα. 500.000 που θα τα βάλουν στην τσέπη τους τα κράτη-μέλη. Είχαμε πει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου να καθοριστούν όλα αυτά, αλλά δεν γίνεται. Το Συμβούλιο ζητάει δε επιταχυμένη διαδικασία. Ο κύριος Ντεπχέ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να κάνω μια διευκρίνηση για αυτό το σημείο των ιδίων πόρων. Δεν είμαι ο μόνος εισηγητή, είμαστε δύο, είμαστε συνεισηγητέ δηλαδή. Από το ΕΛΚ είναι ο κύριο Λεβαντόφσκι συνεισηγητή και λυπάται που δεν μπορεί να είναι απόψε εδώ, αλλά έχουμε διαβουλευθεί οι δυο μας. Και εγώ είμαι λοιπόν ο δεύτερος συνεισηγητής. Ποιο είναι το πρόβλημα. Κάθε χρόνο πριν την 1η Δεκεμβρίου γίνεται ένας επανυπολογισμός και μια επαναπροσαρμογή του ΦΠΑ και των άμεσων ε, εισφορών από τα κράτη-μέλη στην Ένωση, είναι ήδη οι δηλαδή. Αυτή είπατε ότι μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό για φέτος, ε, για κάποιες χώρες συγκεκριμένα, υπήρχαν ε, κάποιες διαφορές, κάποιες επιφυλάξεις, πάντως μετά από μακρές διαπραγματεύσεις επετεύχθη συμφωνία. Το ποσό λοιπόν είναι σημαντικό για κάποιες χώρες τουλάχιστον. Μία εξ αυτών δεν θα την κατονομάσω, αλλά όλη την έχετε στο μυαλό σας φαντάζομαι. Το έκανε μεγάλη ιστορία το όλο θέμα, είπε ότι είναι σκάνδαλο, δεν θα πληρώσει. Κάποιοι μέλη του Συμβουλίου, και θα το πω, το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν, το λέω. Δεν είναι η μόνη χώρα ε, που φύγεται από την αναπροσαρμογή, θα πρέπει δηλαδή να πληρώσει επιπρόσθετα ποσά. Υπάρχει και η Ολλανδία που πρέπει να πληρώσει, υπάρχει η Ιταλία και δυστυχώς και κάποιες άλλες χώρες που είναι σε μια σχετικά λεπτή κατάσταση και αυτό τους έλειπε. Το Συμβούλιο πάντως συμφώνησε επί μία τροποποίησης ε, προς τον κανονισμό 1150 κάθετος 2000 το είπατε και στην τελευταία συνάντηση το συζήτησαν αυτό το θέμα. Τι σημαίνει αυτή η τροποποίηση. Δηλαδή, όταν ζητηθούν ε, σημαντικές εισφορές από κάποια κράτη και υπερβαίνουν είτε για όλα είτε για κάποια από αυτά ένα σημαντικό κατόφλι, υπάρχει δυνατότητα καταβολής ε, με δόσεις αν θέλετε. Αυτό να γίνει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Κάμερον δεν χρειάζεται να πληρώσει τα τρία δις αν δεν εγκριθεί το ε, έκτο σχέδιο ή τέλο πάντων αν εγκριθεί το έκτο ε, σχέδιο διευθυντικού θα είναι άλλο το ποσό. Δεν χρειάζεται να τα πληρώσει όλα το Δεκέμβριο, αλλά μπορεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 να τα πληρώσει. Υπάρχει πρόταση τώρα της Κομισιόν για την τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Η Κομισιόν ε, επέδειξε πιο πολύ επιμέλεια από τη δέουσα επιμέλεια, θα έλεγα, θετικό στην προκειμένη περίπτωση που έδειξε τέτοιο ζήλο. που ε, πόνισε λοιπόν μια πρόταση κατε, κατέτοιμα του Συμβουλίου. Τώρα το Κοινοβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει, να δώσει την άποψή του και το Συμβούλιο μπορεί να κάνει τι θέλει αυτή τη γνωμοδότηση. Και το ελεγκτικό θα γνωμοδοτήσει και το Συμβούλιο θέλει να δώσουμε κατεπηγόντως τη γνώμη μας. Δηλαδή να αποφανθούμε, να γνωμοδοτήσουμε, θα αντιλάβει, θα αντιλάβει υπόψη, κάνει ό,τι θέλει το Συμβούλιο. Θέλει όμως αυτό να γίνει στην Ολομέλεια του τέλους του Νοεμβρίου. Πρέπει να έχουμε λοιπόν να αποφανθεί στο Στρασβούργο για αυτό τον κανονισμό. Και ο κύριος Λεβαντόφσκι και πολλοί άλλοι πιστεύω συνάδελφοι. Τέλο πάντων αυτό έχω ε, νομίζω αντιληφθεί μετά τη συνεδρία των συντονιστών το πρωί. Συμφωνούμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να απαντήσουμε με ε, τόσο πολύ βεβαιασμένη, τόσο, πολύ σπευσμένος ε, και κατεπηγόντος. Φυσικά και θα απαντήσουμε, αλλά γιατί να βιαστούμε τόσο πολύ. Ποιο είναι το κατεπήγον για μας είναι να καταλήξουμε συμφωνία με το Συμβούλιο για τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2014 και για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015. Μέχρι στιγμής έχουμε την εντύπωση ότι πιο επίγον θεωρεί το Σύμβουλο να ρυθμίσει το θέμα των εθνικών εισφορών και όχι να αποφασίσει για τον προϋπολογισμό. Γιατί γενικά δεν έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει σε μια κοινή θέση που να είναι μια αποδεκτή θέση διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο. Ούτε για τους διορθωτικούς του 2014, ούτε για τον προϋπολογισμό, για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2015. Πρόταση λοιπόν και θα ήθελα να την επιβεβαιώσουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Όχι από εκδικητικότητα, αλλά γιατί αλλού βάζουμε εμείς το κατεπήγον. Πρότασή μου λοιπόν είναι να μην εγκρίνουμε το αίτημα κατεπήγοντος του Συμβουλίου, να εξεταστεί δηλαδή κατεπηγόντως αυτή η πρόταση. Να απορρίψουμε αυτό το αίτημα. Και νομίζω ότι πρέπει να επιδείξουμε την ίδια ομοφωνία για αυτό το θέμα, με την ομοφωνία που δείξαμε μέχρι τώρα σε όλε τι διαπραγματεύσει μα με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ναι, και αν είναι αναδρομικό, γιατί πια τέτοια σπουδή. Γιατί τέτοια βιασύνη. Αυτό θα έχει αναδρομική ισχύ ούτως ή άλλως. Κύριος Φερναντές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εκεί που βλέπω εγώ να υπάρχει επίγον χαρακτήρα είναι να ξεπληρωθούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Επομένω να εγκριθούν οι διορθωτικοί προπολογισμοί που εδώ και τόσο καιρό βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιο αρνείται να λάβει θέση. Μιλούμε εδώ τώρα για ένα κανονισμό που δεν ε, ε, φέρνει τίποτα το νέο. Δηλαδή μιλούμε για ένα πρόβλημα το οποίο πάλι είναι πρόβλημα του Συμβουλίου. Ποιο ενέκρινε τον κανονισμό για τους ίδιου πόρους, το Συμβούλιο. Ποιο έδωσε τα στατιστικά δεδομένα για την άμεση συνεισφορά των ε, χωρών μελών από τον προπολογισμό του σύμφωνα με το ΑΕΠ, πάλι το Συμβούλιο. Δεν υπάρχει, δεν βλέπω να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος κατεπήγον χαρακτήρας. Είναι αλήθεια το, συμβούλιο, ο, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο δείχνει πάντα καλή θέληση και επιθυμεί να βοηθήσει το Συμβούλιο για να επιλύσει τις δυσκολίες, να ξεπεράσει τις αδυναμίες. Τώρα όμως υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ των διορθωτικών προϋπολογισμών και τούτο εδώ. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε μέσα σε μια λογική προθεσμία να λύσουμε το πρόβλημα. Όμω το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι είναι κατεπήγον το θέμα των ανεξόφλητων λογαριασμών. Και λένε επίσης ότι αυτό που θα ψηφιστεί θα έχει αναδρομική ισχύ. Μα αυτό αποδείχνει απλά την ανικανότητα του Συμβουλίου να λάβει αποφάσεις πραγματικά σε επίγουσες περιπτώσεις για την Ευρώπη για να ξεπλωθούν λογαριασμοί που έχουν συσσωρεύσει μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει νέοι και ούτω καθεξής. Η κυρία Γκάρδια θα βάλει. Δεν έχω πολλά να προσθέσω μετά από την ε, πολύ πλήρη εξήγηση που έδωσε ο κ. Ντεπρέ. Άλλωστε, συμφωνώ και με τον κύριο Φερνάντες, μπορείτε να υπολογίζετε με τη στήριξή μας των σοσιαλιστών και δημοκρατών διότι και για μας προέχει η εξόφληση των λογαριασμών και να υπάρξει πραγματικός γνήσιος προϋπολογισμός για το 2015. Πραγματικά μας απογοήτευσε ο τρόπος με τον οποίο το Συμβούλιο μπόρεσε να συμφωνήσει πολύ γρήγορα σε αυτά που το ενδιαφέρουν και αδυνα... αδυνατεί να καταλήξει σε μια θέση για τα ζητήματα που επεξεργαζόμαστε εδώ. Ο Πρόεδρος, κύριε Ντεπρέ. Βλέπετε λοιπόν, ακούτε τις απόψεις των συναδέλφων. Μάλιστα, το ακούω. Αν είναι διστακτικέ κάποιε άλλε πολιτικέ ομάδε, ωστόσο θα ήθελα να το ακούσω. Μπορώ να υποθέσω ότι υπάρχει γενική συνένεση μεταξύ μας για το θέμα αυτό. Καλά λοιπόν. Σας ευχαριστώ όλε και όλους. Θα υποκριθώ στην θέλησή σας. Τώρα έχουμε ορισμένα θέματα για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κινητοποιείται μετά από ατύχημα. Μετά από το ατύχημα. εισαγωγικών, δηλαδή το κλείσιμο της επιχείρησης και την απώλεια των θέσεων εργασίας. Έχουμε μια πρώτη έκθεση για την επιχείρηση Whirlpool στην Ιταλία με εισηγητή τον κύριο Βιώτη. Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Αφορά αυτή τη φορά την επιχείρηση Whirlpool στην Βόρειο Ιταλία. Είναι οίκος που κατασκευάζει οικιακές συσκευές και τώρα περιορίζει τις δραστηριότητε του σε λίγες έδρες. Αυτό οδηγεί σε απολύσεις 200 περίπου εργαζόμενους απολύουν στην ε, περιοχή Τρέντο η Ιταλική κυβέρνηση ζητεί 1,8 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Προσαρμογής που ανέρχεται σε 60 περίπου του συνολικού ποσού που δίνεται ως στήριξη στους απολυόμενους εργαζόμενους. Υπάρχει εδώ ένας στάνταρτ μορφότυπος για τις αιτήσει αυτές Η Τετάρτη 12 η είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για να ψηφιστεί μετά στην επόμενη Ολομέλεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αυτά ήταν όλα. Και όποιο επιθυμεί να λάβει το λόγο για την έκθεση του κυρίου Βιώτη, κανένα σχόλιο. Η επόμενη έκθεση, εργοστάσιο της Fiat στην Πολωνία, με εισηγητή τον κύριο Όλμπριχτ. Θα μιλήσω πολωνικά κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Το αίτημα κατατέθηκε από την Πολωνία τον Ιούλιο του 2013. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εξέτασή της διήρκεσε πάνω από ένα χρόνο. Ένα χρόνο και τρεις μήνες μάλιστα. Αυτό μου φαίνεται πολύ μακρά περίοδος, υπερβολική. Πρόκειται για συλλογικές απολύσεις στην Fiat στο Τίσι στην Πολωνία. 1450 εργαζόμενοι. Και σε αυτά προστίθενται 250 προμηθευτές και άλλοι υπεργολάβοι. Το αίτημά μας λοιπόν αφορά πάνω από χίλια άτομα και αφορούσε ποσά χιλιάδων ευρώ. 50% δηλαδή του προγράμματος που έρχεται σε ύψος 2,5 εκατομμυρίων. Θα ήθελα να τονίσω ότι η επαγγελματική τους εκπαίδευση α, είχε αρχίσει και είχαν αρχίσει να οργανώνονται εργαστήρια το πρόγραμμα λοιπόν άρχισε να εφαρμόζεται και τα έξοδα καλύφθηκαν από ποσά που διέθεσε η πολωνική κυβέρνηση που αποφάσισε να μην περιμένει αλλά να αρχίσει την εφαρμογή πριν από τις πληρωμές. Πρόκειται λοιπόν για το θέμα της αποζημίωσης τώρα των δαπανών που έκανε η πολωνική κυβέρνηση. Όλες οι δραστηριότητες που αναλήφθηκαν πέτυχαν και σήμερα χρειάζεται να αποζημιωθεί η πολωνική κυβέρνηση. Μιλάμε για 560.000 ευρώ. Υπάρχει όμως ακόμα μια αμφιβολία. Γιατί η διαδικασία αυτή επαλήθευσης διήρκεσε ένα χρόνο. Γιατί εδώ πρόκειται για κατεπήγον θέμα. Άρα η κινητοποίηση των ποσών θα έπρεπε να είναι ταχύτατη. Η ψηφοφορία θα γίνει το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λίγη στις 4 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα και στις 11 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Στην Ολομέλεια το θέμα θα πάει το Δεκέμβριο επίσης. Ποιος θέλει να εκφραστεί επ' αυτής της έκθεσης του κυρίου Όλμπριχτ, κανείς. Τότε περνάμε στην επόμενη που αφορά την Air Η συγητής είναι ο κύριος Ζάνη. Ευχαριστώ. Στις 11 Νοεμβρίου η Κομισιόν ενέκρινε μία πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για να ενισχύσει τη Γαλλία, για να ενισχύσει δηλαδή τους απολυμένους εργαζόμενους στις αερομεταφορές, ιδιαίτερα την Ερφράνς ΚΑΕΛΕΜ, τη σύμπραξη αυτή. Το ποσό που ζητήθηκε είναι σημαντικό, υψηλό, 26 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθεί το 50% του σχεδίου αναδιάρθρωσης για τους εργαζόμενους αυτούς. Είναι ψηλό το ποσό γιατί ακριβώς είναι πολύ ψηλός και ο αριθμός των απολυμένων. 3.900. 3.860 ακριβέστερα. Απολυμένοι από την 1η Ιουλίου 13 μέχρι 31 Οκτωβρίου 13 έγιναν και άλλες απολύσεις στη συνέχεια στα ίδια πλαίσια. Όπως λοιπόν με την προηγούμενη περίπτωση εδώ η γαλλική κυβέρνηση ήδη είχε αρχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα διάρθρωσης, αναλήφθηκαν προγράμματα δηλαδή στήριξης των εργαζομένων αυτών και τώρα ζητιέται αποζημίωσή τους της δαπάνης των ποσών από την γαλλική κυβέρνηση. Η κατάσταση των αερομεταφορών και των συγκοινωνιών στην Ευρώπη είναι σοβαρή έχει πληγεί πολύ από την κρίση ο τομέας και δύο λόγους για αυτές τις απολύσεις ότι μειώθηκε η δραστηριότητα των μεγάλων αεροπορικών εταιριών αυτό είναι ένα στοιχείο και έπειτα ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση της δραστηριότητας στον Περσικό κόλπο αεροπορικών εταιριών από τον Περσικό κόλπο Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι και, ότι αυξήθηκε πολύ και το κόστος των καυσίμων. Από το 2008 οι τιμές αυξήθηκαν και άρα και το κόστος γινόταν όλο και βαρύτερο για τον προπολογισμό των αεροπορικών εταιριών. Η διορία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, στις 11 ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και ολομέλεια τον Δεκέμβριο επίσης. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης εισηγητής Κύριος Ντινανό. Ναι, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την ανάλυση του συναδέλφου πράγματι Έχουμε μια διαδικασία παγκοσμιοποίησης ε, που δεν αφορά μόνο εξοπλισμό, τεχνολογίες αλλά και υπηρεσίες. Ε, ορίστε ένα σοτανό παράδειγμα, αν μπορώ να το πω έτσι, παγκοσμιοποίησης όπου έχουμε εταιρείε που εξοπλίζονται από τον κόλπο κυρίως, αλλά και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πλήττονται από τον ανταγωνισμό αυτό η γαλλική κυβέρνηση δεν έκανε κατάχρηση της διαδικασίας, πιστεύω. Εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτό που είπε ο κύριος Τζάν, πρόεδρος. Μάλιστα, πολλοί θέλουν το λόγο. Κοιτάξτε, καταρχήν συμφωνούμε με την κινητοποίηση του Ταμείου. Έχω μια ερώτηση, αν είναι και εκπρόσωπος της Κομισιόν πάρω οι ε, νόσεις των εργαζομένων και τα συνδικάτα έχουν ε, γνωμοδοτήσει, ζητήθηκε η γνώμη τους, γιατί μας ανησυχεί πάρα πολύ. Μπορεί να έγιναν οι αιτήσεις στο πλαίσιο το νομικό, ε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και άμεση συμμετοχή των εργαζομένων και των συνδικαλιστών. Είναι κεντρικό σημείο αυτό. Έχετε να μου δώσετε κάποια διευκρίνηση από αυτού παρακαλώ. Ή ο εισηγητής ή η Κομισιόν, πρόεδρος. Κυρία Βάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και μέλος της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Απασχόλησης. Και για την περίπτωση αυτή, αυτή η περίπτωση ήταν κάπως πιο αμφιλεγόμενη. Όχι επειδή δεν είναι ορθά θεμελιωμένη, αλλά είναι σωστό που άλλαξαν οι κανόνες και γι' αυτό το λέω. Διότι η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από ένα κανόνα που δεν υπήρχε ακόμα το 35% των άμεσων επιδοτήσεων. Και επομένω υπάρχει μια δυσαναλογία ανάμεσα στα μέτρα που προβλέπει το Ταμείο, δηλαδή ενεργά μέτρα αγοράς εργασίας για την επανένταξη των εργαζόμενων. Εδώ μιλούμε για περισσότερες direct allowances, 70% λιγότερο. Και γι' αυτό εμείς βέβαια ασφαλώς υποστηρίζουμε και επιδοτήσεις για εργαζόμενους, αλλά υπό τους νέους κανόνες δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει τέτοια αίτηση. Λοιπόν, στο μέλλον, υπό τους νέους κανόνες που ισχύουν, τέτοιου είδους αιτήσει δεν θα μπορούν να εγκρίνονται. Ashworth. Έχω μια περιέργεια για το θέμα αυτό. Βλέπω ότι εδώ ως λόγοι αναφέρεται ο ανταγωνισμός από τρεις αεροπορικές εταιρείε του, κόλπου, του περσικού κόλπου, καθώς και οι πολύ υψηλές τιμές ε, των καυσίμων. Γιατί δεν ισχύουν αυτά και για τη Λουφτχάνσα, για παράδειγμα. 26 εκατομμύρια είναι πολλά λεφτά που πάνε να ρίξουν τώρα στον κλάδο. Δεν θα έπρεπε να δοθεί ε, αποζημίωση και σε όλες τις ε, άλλε αεροπορικέ εταιρείε για παρόμοιους λόγου, για παράδειγμα στη Λουφθάνσα Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι πρόκειται απλώ για ένα μέτρο στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Βεβαίω, δεν είναι αυτή η αρχική πρόθεση. Ούτε είμαι αντίθετο, έχω κάθε κατανόηση για του ανθρώπου που έχασαν τις δουλειέ τους. Αλλά χρειάζεται να επανέλθουμε στους αρχικούς κανόνες της ε, λειτουργία του Ταμείου Προσαρμογή και Παγκοσμιοποίηση για να μην υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ο κ. Φερνάντες. Πολύ σύντομα. Για το θέμα του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, να μην λησμονούμε ότι πρόκειται για συμπληρωματικό ταμείο. Συμπληρώνει άλλα ταμεία, ιδίως το Ταμείο Συνοχής. Ο ρόλος του είναι να ενισχύσει τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις δράσεις των χωρών μελών υπάρχει το Ταμείο, εμείς ερχόμαστε να κρίνουμε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Υποθέσουμε μια χώρα μέλος, καταθέτει μια αίτηση και μια άλλη χώρα μέλος θα είχε δυνατότητα ίσως να κάνει παρόμοια αίτηση με παρόμοιους όρους και δεν το πράττει. Ε, δεν μπορούμε τότε να έρθουμε να επικρίνουμε ή να απορρίψουμε την υπόθεση που εκκρεμεί μόνο για το λόγο αυτό, επειδή οι άλλες χώρες μέλη θα είχαν την ίδια δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις αλλά δεν το έκαναν. Οι κανόνες είναι σαφείς. Και εδώ εμεί καλούμεθα να αναπτύξουμε επιχειρηματολογία για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα. Αν άλλε χώρε υποβάλλουν παρόμοιε αιτήσει, τότε θα ισχύσουν τα ίδια κριτήρια. Προβλέπεται μια διαδικασία. Η αίτηση οφείλει να υποβληθεί σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο κανονισμός και ούτω Αλλά δεν είναι δική μας υπόθεση να ελέγξουμε αν άλλες χώρες έχουν παρόμοια προβλήματα, γιατί και αυτές οι άλλες χώρες μπορούν να υποβάλουν τελειετήσεις αν θέλουν. Ο κ. Να απαντήσω ευχαρίστω στον κύριο Άσχουαρθ. Αν η Λουφτχάνς αντιμετώπιζε δυσκολίες, θα μπορούσαν οι αρμόδιες αρχές να υποβάλουν σχετική αίτηση, αλλά δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες το να ενισχύσει κανείς τους απολυμμένους εργαζόμενους, αυτό ωφελεί τους εργαζόμενους, δεν ωφελεί τις επιχειρήσεις, επομένως δεν είναι στρέβλος του ανταγωνισμού στη Γερμανία. Οι πιλότοι έχουν ιδρύσει επαγγελματικό σωματείο που απεργεί για να αλλάξουν οι συνθήκες εργασίας. Εάν καταλήξουμε σε μια υπόθεση όπου η Λουφθάνσα θα είναι αναγκασμένη να απολύσει εργαζόμενους, αυτό θα έχει σχέση βεβαίως με την πολιτική της Λουφθάνσα, όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, συνδρομή στου απολυμμένου εργαζόμενου, αυτό μπορεί να είναι το καθήκον του Ταμείου πράγματι. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια καθόλου πολιτικά ορθή παρατήρηση ε, έχουμε τους πιλότους της Air France που απεργούν. Δεν κοστίζει αυτό πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων, ε, μήπως φταίει το έχουμε πουλήσει πολλά Airbus σε αυτές τις αεροπορικές εταιρείε του κόλπου και έχουμε τώρα αυτό τον ανταγωνισμό. Γιατί αν αγοράζουν τα καλύτερα αεροσκάφη Airbus οι εταιρείε ε, του κόλπου και πετούν με υφιστάμενο προσωπικό που έχει τελείως διαφορετικό καθεστώς ε, από το ευρωπαϊκό πλήρωμα δεν είμαστε εδώ στο επίκεντρο τη όλη προβληματική για την παγκοσμιοποίηση, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον αυτό το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να παρεμβαίνει όταν δεν γίνεται τίποτα πια, γιατί έχουν χαθεί θέσει εργασία. Ή εάν μήπω θα μπορούσε να παρεμβαίνει με προσπάθειε των κρατών για την εφαρμογή διορθωτικών μεταρρυθμίσεων, ανάκτηση τη ανταγωνιστικότητα και πρόληψη των απολύσεων. Τι είναι αυτό το ταμείο, δηλαδή αφού ε, έχει σπάσει κάτι πάμε να το κολλήσουμε εκ των υστέρων. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς ε, τι προσφέρει αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην ε, παγκοσμιοποίηση. Ούτε τις πρώτες βοήθειες. Η ατροδικαστική έρευνα είναι αυτό. Νεκροτομία κάνει, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πώς θα αποφύγουμε τις απολύσεις. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Άσχουερθ. Αν τολμώ, κύριε Πρόεδρε, να προτείνω, στην περίπτωση βιομηχανιών στην Ευρώπη που έχουν εξαφανιστεί εντελώ ή μετακατασταθεί εξωχώρη ή ε, εξαφανίστηκαν από ε, το βάρος του παγκόσμιου ανταγωνισμού, το καταλαβαίνω. Υπάρχουν ολόκληρες κοινωνίες ε, που βασίζονταν στα θρακοριχεία και μπορεί να έχουν υποστεί μεγάλα πληγματά και έχω απόλυτη συμπάθεια και κατανόηση. Εδώ τώρα μιλάμε για την ε, ικανότητα που έχουν μεγάλες εταιρείες να προσαρμοστούν, να λάβουν ε, τα διοικητικά του συμβούλια ε, τις αποφάσεις τους για να μπορέσουν να αντέξουν στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Κάποιες ε, εταιρείες το καταφέρνουν, κάποιες άλλες δεν το καταφέρνουν. Γιατί θέτω εγώ αυτό το ερώτημα. Εμείς γιατί θέλουμε εδώ να αποζημιώσουμε μια εταιρεία που ίσως καθυστέρησε πάρα πολύ να αντιμετωπίσει από πλευράς δίκαισης το λέω την κρίση και τον ανταγωνισμό συγκεκριμένα. Γιατί η Λουφτχάνσα έκανε τις σωστούς ε, διαγωνισμούς ε, και τη δίκηση αντέδρασε σωστά και απέφυγε το πρόβλημα. Ε, και λυπηρό είναι το ότι στην περίπτωση της Air France δεν έγινε κάτι τέτοιο και έχασαν δουλειά οι άνθρωποι και τους λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έλαβε η εταιρεία τις κατάλληλες αποφάσεις σε επίπεδο διοίκησης. Άρα δεν ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Mais récemment, c'est parce que la compagnie... Η εταιρεία είχε κάνει μια πρόταση <coughs> για να προσαρμοστεί στον ανταγωνισμό με τη δημιουργία μιας θηγατρικής της χαμηλού κόστους και αυτό έδωσε έναυσμα στην απεργία της οποίας το κόστος ε, είναι πολύ ψηλό, πολύ ψηλότερο και από την επιχορήγηση που ζητιόταν. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαπαιδαγωγήσουμε τον κόσμο για τις διαρθρωτικές προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ναι, εδώ είναι δύο προβλήματα κύριε Πρόεδρε. Το ένα είναι οι απολύσει των εργαζομένων που πρέπει να βοηθήσουμε και είναι και το θέμα της εκθέσης αυτής. Και το δεύτερο είναι το παραπάνω για την παγκοσμιοποίηση. Η κυρία Χάουταλα. Με χαίρομαι που γίνεται η συζήτηση αυτή, λέει η κυρία Χάουταλα, γιατί εγώ παρακολουθώ την κατάσταση των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών γιατί και στη φιλανδική κυβέρνηση ήμουν αρμόδια για κρατικές επιχειρήσεις και είδα και τι έπαθε καημένη η Finnair που το κράτος ήταν μέτοχος κατά 66%. Όλες αυτές σιγά σιγά οι επιχειρήσεις πτώχευσαν. Και κύριε Πρόεδρε νομίζω έχετε δίκιο όταν θέτετε το θεμελιώδες ερώτημα πώς μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει καλύτερα την προσαρμογή των αεροπορικών εταιριών στην παγκοσμιοποίηση όπου οι φτηνές εταιρείε αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Και οι συνάδελφοι που τόνισαν την έλλειψη ηγετικών ικανοτήτων των ε, διευθυνόντων ε, των, επιχειρήσεων, πράγματι έχουν δίκιο. Ορισμένες επιχειρήσεις τα πήγαν πολύ καλύτερα από άλλες. Και για να ε, έρθουν και σε διαβουλεύσεις και με οργανώσεις των πιλότων ή του προσωπικού καμπίνας ή του προσωπικού εδάφους κτλ. Η SAS για παράδειγμα τα κατάφερε πολύ καλά, πολύ καλά διότι έφτασε κοντά στην πτώχευση πριν από δύο χρόνια και βγήκε και είπε αυτή είναι η τελευταία μας, η στάτη μας ελπίδα θα πούμε ότι όλοι το προσωπικό από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο θα μειώσει κατά 20% τις απολαβές του. Και συμφώνησαν. Υπάρχουν λοιπόν και άλλες πρακτικές καλύτερες και άλλες βέβαια χειρότερες. Τέλος, ο κύριος Πρέζα για να μας πει πώς λειτουργήσε, πώς αντέδρασε η Κομισιόν, γιατί και αν έχουν γίνει διαβουλεύσεις με το προσωπικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στην Αγγλική. Για τις καθυστερήσεις των πολωνικών αποζημιώσεων Πράγματι πέρασε πολύ καιρό για τη διεκπαιρέωση του αιτήματο, αλλά ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες και δεν δόθηκαν παρά τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να δείτε πώς αντέδρασε η Κομισιόν. Τώρα για το θέμα του κατά πόσον τα συνδικάτα έτυχαν διαβούλευση στην περίπτωση της Air France. Πράγματι έτυχαν και οι προτινόμενοι δέσμοι σε συνδυασμό, σε συμφωνία με τους εκπροσώπους τους έγινε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν ήταν κρατικές επιχορηγήσεις. Η Air πρέπει να αντιμετωπίσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ως προς τις απολύσεις και δεν χρηματοδοτήθηκαν όλα αυτά από, το διαρθρωτικό, από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ήταν μια στήριξη προς τους απολυμένους ώστε να βοηθηθούν να βρουν κάποια άλλη εναλλακτική θέση εργασίας. Εδώ Έρχομαι λοιπόν στο θέμα που συχνά επαναλαμβάνεται. Ποιος είναι ο ρόλος του Ταμείου και πώς θα μπορούσαν να προβλεφθούν όλα αυτά, να προληφθούν. Στον ενωσιακό προϋπολογισμό υπάρχουν εργαλεία που αφορούν τα διαρθρωτικά προβλήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν πιο μακροπρόθεσμα τις συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης καθώς και ανταγωνιστικότητα στην ενωσιακή οικονομία στο σύνολό της. Μάλιστα η Ένωση στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν αντικαθιστά εθνικά προγράμματα. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια για τους εργαζόμενους. Και τέλος, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα από κράτος μέλος για να κινητοποιηθεί το EGF, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία είναι αυτή η συζήτηση. Οργανώνουμε και σεμινάριο επ' αυτού τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. με τα μέσα που μας διαθέτει η διαδικασία του προπολογισμού, αλλά είναι ολόκληρο θέμα χωριστό η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Βάνα για την περίπτωση Οδυσσέως Φωκά στην Ελλάδα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε σύγκριση... Μισό λεπτό διακόπτη Πρόεδρος. Με συγχωρείτε κύριε Βάνα. Η έκθεση μας ήρθε μόλις χθες το βράδυ λόγω ασθενείας του αρμοδίου προσώπου στη γραμματεία. Και βεβαίω μα έχουν δυσκολέψει και όλε αυτέ οι εργασίε για τον προπολογισμό. Ήταν λοιπόν αρκετά καθυστερημένη η διαβίβαση τη εκθέσεως. Έχετε το υπόψη σα αυτό. Μάλιστα, σα ευχαριστώ. Δεν άκουσα μέσω τι μου είπατε, γι' αυτό συνέχισα να μιλώ σε σύγκριση με την προηγούμενη υπόθεση είναι μικρότερη τούτη εδώ. Πρόκειται από την Ελλάδα, πρόκειται για την επιχείρηση Οδυσσεύς Φωκάς του λιανικού εμπορίου είναι αυτό. Μεγάλος λιανέμπορος, ο οποίος λόγω της κρίσης, λόγω των επιπτώσεων της κρίσης, της μείωσης δηλαδή της συζήτηση και της σημαντικής πτώσης του τζίρου εργασιών του, αναγκάστηκε να απολύσει 800 εργαζόμενους. ζητήθηκαν χρήματα για 551, έχουν ε, απορροφηθεί κάποια χρήματα, πρόκειται για 6 εκατομμύρια ευρώ που αποτελούν το 60% της συνολικού ποσού επενδύσεως που προβλέπουν οι ελληνικές αρχές για ενεργά μέτρα για την επανένταξη των εργαζόμενων. Ένα θετικό στοιχείο εδώ είναι ότι εδώ μπαίνουν και κάποια χρήματα από την εγγύηση των νέων. 500 νέοι δηλαδή λαμβάνουν υποστήριξη για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόκειται για 89% γυναίκες, διότι γνωρίζουμε ότι ιδίω στο ελληνικό εμπόριο εργάζονται γυναίκες. Επίσης θετικό είναι το πόσο γρήγορα αντέδρασαν οι ελληνικές αρχές. Η αίτηση από την πλευρά της Ελλάδος έγινε στις 29 Εβδόμου. Έδωσαν κάποια πρώτα χρήματα οι ελληνικές αρχές για να βοηθήσουν γρήγορα από τον Οκτώβριο ήδη τους εργαζόμενους. Στις 11 Νοεμβρίου ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η υπόθεση δηλαδή εμπίπτει στους κανόνες του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και η διαδικασία εξελίσσεται μέχρι τις 4 12 είναι η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών. Στις 11-12 η απόφαση εδώ στην Επιτροπή και μετά εγκρίνεται στην Ολομέλεια το Δεκέμβρη. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Άρα, περνάμε στην ψηφοφορία. Πρόκειται για προηγούμενες ε, κινητοποίησεις τις οποίες πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Πρώτη. Φιλανδία, Ράουμα, Σαβαμό εισηγητής, έχετε λάβει τις τροπολογίες. Στην παράγραφο 3 έχουμε την τροπολογία 1. Είμαστε εντάξει με αυτήν. Παράγραφος 4 Τροπολογία του εισηγητή. Θέλει το λόγο για τις τροπολογίες που πρότεινε μήπως εισηγητής. Α, δεν ακούω τι μου λέτε, αλλά... Α, τα έχει πει, λέτε, μάλιστα. Και είναι υπέρ. Είναι υπέρ των τροπολογιών. Πώς προτείνει, μάλιστα. Ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Κατά. Δεν βλέπω. Ούτε αποχές βλέπω. Παράγραφος 5. Τοπολογία 2. Ο εισηκτής υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Τρεις βλέπω. Αποχές δεν υπάρχουν. Παράγραφος 11. Τοπολογία 3. Ο εισηγητής υπέρ. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Νομίζω σκόστε όλοι τα χέρια. Άρα δεν υπάρχει κανείς κατά, ούτε και απέχει κάποιος. Παράγραφος 12, το 5, ποιοι είναι υπέρ, είναι υπέρ ο εισηγητής. Κατά, αποχές δεν βλέπω, τροπολογία 6, ο εισηγητής υπέρ, ψήφι υπέρ. Κατά, 3 αποχές όχι. Τροπολογία 7. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω. Ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε τώρα επί του συνόλου του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. εγκρίνεται 19 υπέρ 3 κατά καμία αποχή. Έκθεση Γκάντ, Γαλλία. Η συγκίτρια κυρία την Τενμάκη. Έχετε κυρία μου παρατηρήσεις για τις τροπολογίες. Όχι. Άρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Είναι αρνητική άποψη της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Είναι υπέρ Ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, για την παράγραφο 6. Ψηφίσατε όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η παράγραφος 6. 16 υπέρ 9 κατά. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω την κάρτα μου μαζί. Θα σηκώνω το χέρι αν μπορείτε παρακαλώ να με υπολογίζετε και εμένα. Μα είστε αναπληρωματικό μέλος. Από πού? Α, καλά, εντάξει. Ήσασταν υπέρ τώρα? Δεν αλλάζει και τίποτα. Ναι, θα είναι απλά 16 προς 10 το αποτέλεσμα. 6 κατά 10 υπέρ. Λοιπόν, οι 16 υπέρ, μάλλον 10 κατά. Για να δω που είμαι γιατί τα έχασα. Παράγραφος 6, τροπολογία 3. Η εισηγήτρια είναι αντίθετη. Ψήφι υπέρ της τροπολογίας 3. Ακούστε, ας περάσουμε κατευθείαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Βάλτε και η μερνητική ψήφο παραπάνω. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ 11 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία. Στην παράγραφο 14α τροπολογία 4. Η συγγήτρια υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 15 Συμπλήρωμα α, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Ο πρόεδρος πρέπει να εννοεί συμβιβαστική α. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, 8 κατά. Εσείς τι είχατε ψηφίσει κατά, ωραία. 18 προς 9, λοιπόν. Τροπολογία 7 στο 15, ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν υπάρχει. Αποχές. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, αλλά καλύπτεται. Πού πάμε καλύπτεται αφού ψηφίσαμε το συμβασμό. Πάμε. Στη 15α νέα. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Η σύγκεντρα είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Η σύγκεντρα είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ουδής. Ούτε και αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Η σύγκεντρα είναι υπέρ. Κατά που ούτε και αποχές. Τροπολογία 12. Η είναι αντίθετη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 16 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 4 αποχές. Εσείς τι ψηφίσατε κύριε, υπέρ, άρα 17 προς 6. Στο 15ε, τροπολογία 13, ποιοι είναι υπέρ. Κατά, τίποτα, κανείς, όλοι υπέρ. 16α τροπολογία 14. Η σύντρα είναι θετική. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Κανείς. Ούτε αποχές. Τροπολογία 15. Ψήφι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές 2. Τροπολογία 15. Το ψηφίσαμε. Α, το ψηφίσαμε. Πού πάμε δηλαδή τώρα. Α, στην ετολική σκέψη ε, α, το recital ε, τροπολογία 1. Υπέρ εισηγητρία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, α, Recital, λειτουργική σκέψη. Δύσκολη εβδομάδα, ε. Πέρα της ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε ονομαστικά, ηλεκτρονικά δηλαδή, όλο το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Μπορέσετε να ψηφίσετε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν με 23 ψήφους υπέρ και 3 κατά. 24 ψήφους υπέρ με τον κύριο εκεί. Τώρα περνάμε στην έκθεση του κ. Φερνάντες. Κύριε Ντεπρέ, πριν δώσω το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Ντεπρέ. Oui, vous la parole avant le vote sur ce rapport. Τι θέλετε το λόγο πριν ψηφίσουμε την έκθεση Φερνάντες. Να μην δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Φερνάντες. Κύριε Φερνάντες δεν έχετε να πείτε κάτι, ωραία. Κύριε Ντεπρέ, εσείς. Κύριε Πρόεδρε, είναι λίγο ιδιόμορφη η ψηφοφορία για την Άλντε. Σκιώδης η συγκητής ο κύριος Στόρβαλς δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν. Και παρά τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει για τον συνάδελφο κύριο Φερνάντες, έκανα κάποιους υπολογισμούς και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό που μας ζητούν να ψηφίσουμε εδώ θα κοστίσει πολλά. Θα στοιχήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τους υπολογισμούς. Ξέρετε ότι πρέπει να δίνει ε, με αντάλλαγμα αλλιευτικές ποσοστώσεις κάποια χρήματα η Ένωση. Για ένα δολάριο, μάλλον για ένα ευρώ που επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνει τη μετρητής, θα έχουμε επιστροφή 40, 45 λεπτών του ευρώ με τα αλλιεύματα. Μας ζήτησε να στηρίξουμε την επιχειρηματολογία, θα ψηφίσουμε περίεργα δηλαδή. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία του 1, που μάλλον θα απορριφθεί και όταν απορριφθεί και εφόσον απορριφθεί θα, πληρώ, θα, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε παρόλα αυτά υπέρ της έκθεσης. Αυτά ε, για να ξέρουμε ε, τελικά τι δεσμεύσεις κάποιες φορές αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και προς στιγμήν αφού είμαστε στην ψηφοφορία δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση. Οι επεξηγήσεις ψήφου γίνονται μετά την ψηφοφορία. Τώρα θα ξαναρχίσουμε συζήτηση, ε, εντάξει, άμα θέλετε, εντάξει. Αλλά μετά να ψηφίσουμε. Υπάρχει και προηγούμενο. Τα ποσά δεν είναι πολύ ψηλά, όλα είναι δικαιολογημένα. Αν θέλουμε να ξαναρχίσουμε συζήτηση, επαναλαμβάνω, ας το κάνουμε. Και Πιστεύω όμως ότι δεν είναι τη στιγμή της ψηφοφορίας η καταλληλότερη στιγμή. Οι επεξηγήσεις ψήφου υπάρχουν, αλλά γίνονται, το λέω για τρίτη φορά, μετά την ψηφοφορία. Ο κύριος Δεπρέ μας είπε ότι δέχεται το κείμενο. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 1 του κυρίου Τόρβαλτς. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα ηλεκτρονικά για το σύνολο του κειμένου που δεν τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Pardon? Άρχεται η ψηφοφορία, είπαμε. Il y en a Μερικοί δεν ψήφισαν. Έληξε. Ψήφισαν όλοι. Λοιπόν, 18 υπέρ, 5 κατά. Περνάμε τώρα στο τμήμα 3 του προπολογισμού 14 με τις μεταφορές. Κύριε Ντεπρέ. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Ντεπρέ. Μια στιγμή να ξαναδώ τα χαρτιά μου εδώ μετά από αυτά που μου είπε ο κύριος Φερνάντες ταράχτηκα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν προβλήματα με τις μεταφορές κύριε Πρόεδρε. Δύο είναι. Οι 36 και οι 38 που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστούν τα ποσά για την εκτέλεση των αποφάσεων που πήραμε για ταμεία στήριξης, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται πια, αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης. προσαρμογής μάλλον στην παγκοσμιοποίηση και αυτές ήταν οι μεταφορές 36 και 38 λοιπόν. Η 39 αφορά πολύ μικρό ποσό 1,2 εκατομμύρια για την European Medicine Agency. Υπάρχουν κονδύλια για τις πληρωμές σε αυτήν την European Medicine Agency που θα ήταν πολύ χρήσιμα να δοθούν ανταυτής στην Eurojust που θα τα χρησιμοποιήσει για μισθούς και συντάξεις. Αποσαφηνίζω ότι η μεταφορά 42 ζητώ να συνεννοηθεί με την κυρία Γκρέσλε η Κομισιόν που ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες αλλά ούτως ή άλλως θα την εγκρίνουμε γιατί προσωπικά εγώ δεν έχω αντιρρήσεις στην επόμενή μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Για την 36 και 38 είναι υπέρ ο εισηγητής. Νομίζω ότι ε, ακολουθούμε και οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν αυτών των μεταφορών οδικών στο χέρι τους. Ευχαριστώ κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Για την 39 θα επανέλθουμε. Α, όχι, είναι και, ε, και για αυτήν υπέρ ο εισηγητής. Λοιπόν, για την 39 υπέρ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Λοιπόν, κυρία Μέγερ, για τα υπόλοιπα τμήματα υπάρχουν επίσης προτάσεις μεταφορών. Για τους άλλους τομείς έχουμε μία μικρή υπόθεση γλωσσικές εκπαιδεύσεις για τους νέους ευρωβουλευτές και λείπουν εκεί 5.000 ευρώ. Και αυτά να εξευρεθούν με κάποια μετακίνηση ε, πόρων μέσα στον προπολογισμό άνευ προβλήματος. Για το ελεγκτικό συνέδριο, τέσσερις μεταφορές, επίσης από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Για λόγους υγιεινής στο εστιατόριό τους πρέπει να αλλάξουν κάποια υλικά Δεύτερο, έχει χαλάσει ένα μηχάνημα εκτύπωσης και πρέπει να αντικατασταθεί. Τρίτο, στον χώρο συνεδριάσεων πρέπει να ε, αντικατασταθούν κάποια μηχανήματα που δεν λειτουργούν. Και τέλος, τα συστήματα πληροφορικής πρέπει να επαναπρογραμματιστούν μετά από τις παραπάνω αλλαγές 50.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, 55.000 ευρώ και 380.000 ευρώ. Συνολικά μέσα στα πλαίσια των προϋπολογισμών, μέσα στα πλαίσια των ε, πόρων που αρμόζουν στα διάφορα, διάφορα θεσμικά όργανα και επομένως από εμά εγκρίνονται. Ποιος θέλει το λόγο, δεν βλέπω κάποιος να θέλει το λόγο. Ποιοι είναι υπέρ των μεταφορών πιστώσεων, παρακαλώ. Νομίζω σχεδόν όλοι ήταν υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποφέ, αποχές, συγγνώμη. Κυρία Χολμάγερη, έχετε πάλι το λόγο για την κτηριακή πολιτική. Τι γίνεται με αυτό το κτίριο στη Λισαβόνα, που είναι νομίζω φαντα... είναι φανταστικό. Εδώ είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεση, θα προσπαθήσω να τα πω σύντομα. Πρόκειται για τον διακόπτη κάποιος. Όχι, όχι, εντάξει πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Παλαιότερα ο οργανισμός αυτός διέθετε κτίριο που το αγόρασε 2,95 εκατομμύρια και χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 2009. Μετά η κρίση χτύπησε και την Πορτογαλία, έπεσαν οι τιμές των ακινήτων και δεν μπόρεσαν τα τελευταία πέντε χρόνια να το πωλήσουν το ακίνητο. Τώρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος προσφέρει τέλος πάντων 2,5 αντί των 2,95 εκατομμύρια. Υπάρχει και προσφορά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μισθώσει το κτίριο για δύο χρόνια και διατίθεται να πληρώσει 80.000 ευρώ μίστομα και να το αυξήσει κιόλα, εγώ πιστεύω ότι είναι σκοπιμότερο να απολυθεί το, το ακίνητο. Δεν είμαστε ε, μεσίτες, δεν είμαστε εμπόρια κινήτων. Καλύτερα να απολυθεί το κτίριο αντί να επιβαρυνθούμε και με έξοδα συντήρησης κλπ. Νομίζω ότι αυτά 2,5 εκατομμύρια είναι ικανοποιητική τιμή εν ώψη και της κρίσεως. Ο οργανισμός θα ε, συγκατοικήσει εντός εισαγωγικών μαζί με άλλο οργανισμό έτσι ώστε θα προκύψουν και κάποιες οικονομίες. Εσείς κύριε Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως προτείνει η κυρία Χολμάγερ, πιστεύω πράγματι και εγώ ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε με το θέμα αυτό. Βέβαια, σε σχέση με την αρχική τιμή, είναι σοβαρή η μείωση. Με βάση τις βασικές ε, εκτιμήσεις, 3,4 ή 3,5 δις, ε, τώρα μιλάμε για 20. Καλό το νέο τέλος πάντων ε, και γίνεται χωρίς την παρέμβαση κάποιου μεσητικού γραφείου. Γιατί αν δει κανεί τι τιμέ, συγγνώμη, μιλάμε για 2,5, όχι για 20. Ε, τα λέω στον ε, συνάδελφο Φερνάντε. επειδή βλέπω να είναι υπερβολικέ απαιτήσει αυτών των οργανισμών, μήπω πρέπει να του τραβήξει τα αυτή λίγο. Ένα-ένα, κύριε Φερνάντε, τώρα. Σα ισοφάρισε ο κύριο Ντεπρέ. Λοιπόν, Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της κυρίας Χολμάγερ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δύο. Άρα είμαστε υπέρ ως Επιτροπή. Προπλωσμό στην πρόταση της κυρίας Χολμάγερ. Άλλα θέματα, διάφορα. Στα διάφορα υπάρχει κάτι όχι. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να συνέλθουμε όλοι από τις αποτυχημένες συνδιαλλαγές.